Η Ισπανία είναι αυτή που είχε στείλει πολεμικά πλοία. Διακόπτει ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι διαδικαστικό. Περνάμε λοιπόν στις ψηφοφορίες για την πρόταση ψηφίσματος, κοινού ψηφίσματος του ΕΛΚ Σοσιαλιστών ΑΛΔΕ, του ΓΚΟΕ, Πρασίνων και Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων ε, ψηφίζουμε για την τροπολογία 18. Il voto è chiuso. Τέλος της ψηφοφορίας πρόταση, ε, αυτό απορρίπτεται. Περνάμε στο αρχικό κείμενο, ονομαστική κλίση, άρχεται. Il voto è chiuso. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφο 7, αρχικό κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. εμποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9, παράγραφος ε, ε τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στο αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφό 11. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Μετά από την παραγραφή 11, τροπολογία 13, ονομαστική κλίση, ε, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Παράγραφος 12, τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 13, τροπολογία 16, ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 17, αρχικό κείμενο, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εκρίνεται. Μετά την παράγραφο 18, τροπολογία 8, ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Περνάμε στο αρχικό κείμενο, ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Εκρίνεται. Μετά την παραγραφή 20, τροπολογία 20, ονομαστική κλίση άρχεται. αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 ονομαστική κλίση άρχεται. Voto è chiuso. Πέρας. Απορρίπτεται. Μετά από την παράγραφο 9, τροπολογία 9, με ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος, απορρίπτεται. Περνάμε στο αρχικό κείμενο της παραγράφου 23. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 24. Αρχικό κείμενο. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 25, αρχικό κείμενο, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 27. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Il voto è chiuso. Εγκρίνεται. Παράγραφος 28. Αρχικό κείμενο. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Il voto è chiuso. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 31. Πρώτο τμήμα. Ε, κατά ε, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Τέλος, εγκρίνεται. Παράγραφος 32. Ορχικό κείμενο. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά από την παράγραφο 35, τροπολογία 15, νομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19, νομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Εκτιμώντα β, αρχικό κείμενο, δύο τα πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας Ι, ε, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση. Πέρας, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας μη. Αρχικό κείμενο. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας νη. Τροπολογία 1 και 5. Ονομαστική κλίση. Άρχεται.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 Τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική κλίση «Άρχεται». Ψηφίζετε όλοι. Πέρασε. Τώρα εγκρίθηκε με 516 ψήφους υπέρ. 133 και 133 ψήφους κατά και 50 αποχές.